Iniziamo, colleghi. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Se non vi sono obiezioni, colleghi, intanto benvenuti a tutti. Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι, πρώτον. Δεύτερον, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Να σας ανακοινώσω και με χαρά επίσης ότι σήμερα έχουμε διερμηνία διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η σημερινή συνεδρίαση ε, μεταδίδεται και μέσω webstream. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών της συνάντησης 31 Ιανουαρίου της περασμένης ε, συνάντησης. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Ξεκινάμε με το σημείο 5. Γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης ε, στο περιβάλλον, για το περιβάλλον μέχρι το 2020. Ζώντας καλά μέσα, ζώντας καλά μέσα στα όρια του πλανήτη μας. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Σάρμπου, εδώ. Θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοζώτησης επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα αυτό είναι το έβδομο πρόγραμμα δράσης από το 1973 και μετά, μετά από μια σειρά διαδοχικών προγραμμάτων πλαίσιων. Ε, αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και εμείς παρέχουμε μια γνωμοδότηση. Δίνω μέσω στο λόγο στην Ντατσάνα και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, ε, τον θυμίζω σε όλους, του συναδέλφου είναι αύριο 5 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Θα εγκρίνουμε την γνωμοδότηση στην Επιτροπή 18-19 Μαρτίου, ενώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφιστεί η γνωμοδότηση 24 Απριλίου. Η κυρία Σάρμπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο αυτό για το θέμα που ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά στόχων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Θέλουμε να υπάρξει μια μετάβαση σε μια αποτελεσματική οικονομία που εκμεταλλεύεται σωστά τους πόρους και έχει μειωμένες εκπομπές για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το φυσικό κεφάλαιο και να διαφυλάξουμε την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Ο κλάδος της γεωργίας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων. Φερρυπίν την αύξηση της ανάγκης σε τρόφιμα, τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και όλο ένα και μεγαλύτερες επιπτώσεις από την θέρμανση του πλανήτη. Βάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο τομέας αυτός είναι υπεύθυνο κατά 9,5% για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Ο κλάδος γεωργίας δηλαδή. Ταυτόχρονα, η γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η δασοπονία, παίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των, ε, της αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα και την διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Το Κοινοβούλιο αναγνώρισε στην θέση του εν ώψη του 2020 ότι η καινοτομία στην γεωργία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τον ε, περιορισμό των εκπομπών και για τον περιορισμό των συνεπειών της παγκόσμιας ε, υπερθέμανσης η γεωργία μας θα πρέπει να παράγει περισσότερα με λιγότερους πόρους, άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ορθολογική χρήση των πόρων αυτών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διορθώσουμε ε, τη διασπάθηση τροφίμων. Πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη και τον ε, σημαντικό ρόλο της γεωργίας και να διασφαλίσουμε ότι τα παρασιτοκτόνα που έχουν αρνητικές ε, επιπτώσεις στη μελισσοκομεία θα απαγορευτούν. Η νέα γεωργική πολιτική θα πρέπει να αποζημιώνει με σωστό τρόπο τους γεωργούς. Τρία είναι τα μέτρα που προτείνονται στην ε, Επιτροπή. Διαφοροποίηση των καλλιεργειών, θέσπιση ε, μόνιμων λιμόνων και χορτονομών και εγγύηση ότι η βιωσιμότητα της γεωργίας. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι οι, γεωργικές, οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η βιολογική γεωργία θα πρέπει να προωθηθούν με πολύ περισσότερο μεγαλύτερο τρόπο διότι ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα υπάρχουν σαφείς, ε, σαφή πλεονεκτήματα και για τους καταναλωτές. Επιπλέον χρειάζεται να προωθήσουμε μια σειρά ε, πιο σύντομες, πιο βραχίες αλυσίδες ε, τροφοδοσίας και να λάβουμε υπόψη τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να έχουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας που, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και στους μικρούς γεωργούς που είναι βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή γεωργία. Κλείνω ευχαριστώντας σας ε, για την προσοχή σας και για τη συμβολή, ε, συμβολή σας. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις τοπολογίες. βέβαια μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Η αντιπρόεδρος Πόλσον πρώτα και κατόπιν η κυρία Κλάς. Κυρία Πόλσον. Ευχαριστώ. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή είναι πιστεύω ε, αγνοεί πιστεύω πλήρως τα θέματα της γεωργίας. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρηθούν αυτοί το μέρος της λύσης. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω μια σειρά από τροπολογίες. διότι υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος, αναμφίβολα. Ε, και έτσι το πιο σημαντικό νομίζω θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η παραγωγή τροφίμων για τον επιστησμό μιας περιοχής. Και αν μας επιτρέπει η παραγωγή να έχουμε ικανοποίηση αυτών των αναγκών, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Μέσα σε έναν κύκλο φυσικό που φαίνεται να έχουμε ξεχάσει. Επίσης, η δασοκομεία ξεπερνά τα απλά όρια του δάσους. Ξέρουμε βεβαίω ότι, ότι τα δάση λειτουργούν και ω αποθετήρε άνθρακα και ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Λυσμονούμε ωστόσο ότι είναι πηγή ανανεώσιμων πόρων το δάσος. Εάν κάποια στιγμή η γη μας αριθμεί 10 δισεκατομμύρια κατοίκους, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο. πολύ περισσότερους σπόρους. Αυτούς τους σπόρους μας τους προσφέρουν τα δάση. Και στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερους σπόρους με τα δάση, με το χαρτί, με όλα τα προϊόντα των δασών. Σας παρακαλώ λοιπόν στην ψηφοφορία ε, να λάβετε υπόψη την αντίρρηση που προβάλλω διότι είναι κέρια σημασίας. Ε, είναι μία πηγή πόρων το δάσος και δεν σχετίζεται μόνο με τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον. Είναι τόσο σημαντικό το δάσος που μας επιτρέπει να έχουμε βιώσιμους φυσικούς πόρους και αυτά που παράγουμε σήμερα με το πετρέλαιο μπορούμε να τα παράξουμε στο μέλλον χάρη στα δάση. E Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Σάμπου για την έκθεση πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο δεν μπορεί βέβαια να αποκοπεί από τη γεωργία όπως και να έχει. Είπε και στην αλφός μόλις τώρα ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη δασοκομεία. Το ίδιο και για τη γεωργία. Πρέπει να δούμε τι ε, πώς βλέπει την ε, γεωργία γενικότερα ο κόσμος. Και θα ήθελα με το πρόγραμμα δράσης να ρωτήσω τα εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν ε, πολλέ αρνητικές παρατηρήσεις και δεν είμαι βεβαία ότι χρειάζεται πράγματι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Καλό είναι να υπάρχουν οι στόχοι, με αυτού θα προχωρήσουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα περιγραφεί αυτός ο, ο, ο που θα φτάσουμε στις επιλογές μας, δεν νομίζω ότι είναι θεόπνευστος. Ίσως ε, υπάρχει περιθώριο στη διάρκεια ενός προγράμματος να γίνουν διορθώσεις και αλλαγή πορείας. Άρα λοιπόν, εάν βλέπουμε ότι ο δρόμος που στρώνουμε χρειάζεται νέο λιθόστρωτο, τότε θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική προσαρμογή. Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού δικαίου στα κράτη-μέλη χρειάζεται βελτίωση, το λέει η Επιτροπή, το λέμε και εμείς βεβαίως και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Και θα πρέπει να ζητήσουμε νέους και πολύ πιο σαφείς περιβαλλοντικούς νόμους με στόχους συγκεκριμένους που θα υλοποιούνται πραγματικά. Ε, κριτική λοιπόν θεώρηση του υφισταμένου δικαίου, της υφισταμένης νομοθεσίας και ε, παρακολούθηση της υλοποίησης και με όλες τις αιτιολογημένες επιφυλάξεις μπορεί κανείς να έχει. Εγώ θα διαφωνήσω προς την κατάληξη και την αρνητική κρίση ή την παραγνώριση ακόμη θα έλεγα κάθε είδους επιτεύγματος ή επιτυχίας. Αυτός ο, τόσο, ο τόνος απεσιοδοξίας που διαπιστώνω ε, νομίζω ότι περιτεύει στο κείμενο γιατί αν έχουμε πάντοτε αρνητική στάση τότε μήπως τελικά το ερώτημα που ακολουθεί, που έπεται είναι τι έχει καταφέρει η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια σε τι χρησιμεύει. Δεν νομίζω ότι θα πείσουμε κανέναν με αυτή την οτροπία, ούτε θα κερδίσουμε τη συμπάθεια κανενός για την περιβαλλοντική μας πολιτική. Πολλά είναι λοιπόν αυτά που έχουν υλοποιηθεί και πρέπει να τα προβάλλουμε. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Εδώ, όποια προβλήματα ενδεχομένω εντοπίζονται, ε, εντοπίζονται στην ε, αδυναμία ή ανεπάρκεια εφαρμογής σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, η ανεπαρκεια εφαρμογή σε επιπεδο κρατων μελων επισης η προστασια των εδαφών της γη. Ε, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της οδηγίας και την προστασία των εδαφών. Έχουμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε ως λύσεις, για, ως νομοθετήματα δηλαδή για την προστασία των εδαφών, φυτοπροστασία, δίκαιο για τα απόβλητα, για τη χρήση των γεών, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποτελούν ένα σύνολο νομοθετικό για την προστασία των εδαφών. Αντίθετα με το είδωρ και τον αέρα, είναι ένα υλικό, ένα στοιχείο που δεν μετακινείται το έδαφος και βεβαίως εδώ ε, κατά πρώτο λόγο αρμόδια για την υλοποίηση και την εισαγωγή αλλά και την υλοποίηση του δικαίου είναι τα κράτη-μέλη και όχι η ευρωπαϊκή διάσταση. Θα πρέπει επίσης ε, να δούμε οι λύσεις που εισάγονται εάν έχουν οικονομική, οικολογική, ε, κοινωνική στήριξη και νόημα και αν τελικά βελτιώνουν την αηφορία των πόρων μας, των φυσικών, την δυνατότητα να καλύψουμε τις ε, ανάγκες μας, δεδομένης και της πάνω ε, και εν τέλει την ανάγκη να παράγεται περισσότερη τροφή για να χορταίνουν οι κάτοικοι του πλανήτη. Υπάρχει ανάγκη για παραγωγή κατά τρόπο βιώσιμο καλών προϊόντων, για διάθεσή του στην αγορά κατά τρόπο σωστό. Και βέβαια εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την, την ε, περιφερειακή διάσταση, δηλαδή πόλεις των προϊόντων στην τοπική τους αγορά, και προβολή των περιφερειακών προϊόντων. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω οι θετικές πτυχές, να μην μιλάμε μόνο αρνητικά δηλαδή, αλλά με περισσότερο θετικό πνεύμα να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, προτάσεις και να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα με θετικό πνεύμα. Πολλά έχουν επιτευχθεί και στους άλλους τομείς, θα σημειώσω. Στην πατρίδα μου, τη Γερμανία, παραδείγματι, από το 90 οι εκπομπές θερμοκηπίου έχουν πέσει κατά 18%, αμμονίας ε, κατά 20%, αζωτούχων επίσης, σε σημαντικό βαθμό έχουν μειωθεί οι εκπομπές αζωτούχων αερίων. Ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να υπογραμμίζουμε τις θετικέ πτυχές. Βεβαίως οτιδήποτε είναι ε, στραβό θα πρέπει να το κοιτάμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να κάνουμε τις σχετικές προσαρμογές. Αλλά έχουμε νομίζω το περιθώριο και τη γνωμοδότηση του, α, της Επιτροπής Γεωργίας να κάλυψουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, Έρικ και μετά Ελίζαμπετ. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης που εξετάζουμε παρουσιάζει τις προκλήσεις ε, της γεωργίας σήμερα για να καλύψει τις ανάγκες ενός πληθυσμού που αυξάνεται με μειώνοντας τους κινδύνους. Ο στόχος είναι να παράγουμε περισσότερο και καλύτερο. Η εισηγήτρια, την οποία ευχαριστώ για την ε, έκθεση, τονίζει ότι, το κοινό, ότι η Γεωργία μπορεί να παίξει έναν θετικό ρόλο. Συμφωνώ με τις ε, απόψεις της ότι ε, η φωτοσύνθεση των φυτών είναι βασικός παράγοντας συγκράτησης του διοξιδίου του άνθρακα. Το κείμενο παρουσιάζει μια σειρά καινοτόμων ιδεών ε, για τη γεωργία με τις οποίες συμφωνώ. Προσθέτω ότι προσθέτει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, και ορισμένα μέτρα του δεύτερου πυλώνα επιτρέπουν θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία. Ταυτόχρονα τονίζει την ε, ανάγκη καταπολέμησης της διασπάθειας. Συμφωνώ με τις προτάσεις της ηγήτριας, θεωρώ ωστόσο ότι δεν είναι επαρκής και μειώνουν τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου όταν όπως είχε ξεκινήσει τονίζοντας ε, τις ανάγκες για την αλλαγή της ΚΑΠ. Μιλώ για μια σειρά εκθέσεων για την ε, κατάσταση της γεωργίας μετά το 2013. Η γεωργική ανάπτυξη όπως ε, ασκείται μετά τον πόλεμο δεν μπορεί να παραμείνει όπως έχει μέσω και μακροπρόθεσμα. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο. Κάποιοι ποδι όπως ε, το νάτριο και ο φωσφόρος ε, χάνονται ή σπανίζουν και ακριβένουν όλο και περισσότερο. Τα χημικά ε, μόρια, χημικά μόρια όλο και πιο σύνθετα ποικίλουν και κοστίζουν όλο και περισσότερο. Η χρήση του ύδατος θέτει όλο ένα και περισσότερα προβλήματα. Η ποιότητα του εδάφους υποβαθμίζεται, η βιοπικιλότητα μειώνεται δραματικά πρέπει να αλλάξουμε όχι ορισμένες πρακτικές αλλά ολόκληρο το μοντέλο παραγωγής σήμερα και θα χρειαστεί να διαλέξουμε. Τούτο μπορεί να γίνει με συστημική προσέγγιση που, που αφορά και τα προβλήματα του εδάφους, του νερού και την ε, μείωση της βιοπικιλότητας. Αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην ε, ε, γεωπονία και την οικολογία, αυτό που αποκαλούμε ε, απαιτεί και αλλαγή του υποδείγματος, του μοντέλου παραγωγής. Η παραγωγικότητα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στην φυσική λειτουργικότητα και όχι σε χημικά στοιχεία. Ε, ο κύκλος του άνθρακα, ο κύκλος του αζότου, ο ρόλος των ε, οργανικών ε, υλών στο έδαφος, η βιολογική ζωή του εδάφους. Και αυτό, δεν, και αυτό περιλαμβάνει και βιολογική γεωργία, αλλά και γεωργία που βρίσκεται μεταξύ της συμβατικής και της και της οικολογικής γεωργίας. Πρέπει να μπορέσουμε να παράσχουμε ε, βιώσιμη γεωργία που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές διαστάσεις μακροπρόθεσμα. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να συνοδεύεται από τεχνολογικές μεταβολές που εξασφαλίζουν την μετάβασή μας σε, τα, σε αυτά τα νέα ε, στοιχεία της γεωργίας. Η μετάβαση αυτή πρέπει να προχωρήσει σταδιακά, αλλά πρέπει να προχωρήσει από σήμερα ήδη. Είναι καιρός η προσέγγιση αυτή είναι μια παγκόσμια προσέγγιση για τα προβλήματα του εδάφους, του νερού, της βιοπικιλότητας και της ρήπανσης. Αυτές οι νέες μορφές γεωργίας θα πρέπει να μπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων διεξόδων και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μέσω της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από τα απορρίμματα, την παραγωγή άγροηλικών και την δημιουργία αυτού που αποκαλούμε πράσινης χημίας. Αυτές οι μορφές γεωργίας ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον και για τους λόγους αυτούς η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να γίνει σε βάθος και είναι αναγκαία. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να μπορούμε να επενδύσουμε στην καινοτομία όπως το προτείνει η πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Καινοτομία που προβλέπεται στο δεύτερο πυλώνα. Χρειάζεται επένδυση στην έρευνα, επένδυση, μεγαλύτερη επένδυση στην συμβουλευτική για μεγαλύτερη βιωσιμότητα στους γεωργούς και ε, όπως το προβλέπει ακριβώς ο οριζόντιος κανονισμός για τις μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας τις γνώσεις και την ικανότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία και μετά ο Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την υποβολή της εκθέσεως. Ήδη οι προλαλήσαντες επεσήμαναν τα κύρια σημεία αλλά και τις θετικές ε, πτυχές της εκθέσεως. Εκεί ιδιαίτερος όπου γίνεται λόγος για, την, ε, για τις μεγάλες πατάλες σε τρόφιμα. Και πιστεύω εδώ ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συζητήσουμε πολύ πιο εντατικά αυτό το θέμα. Και μένα η αρνητική προσέγγιση που διαπιστώνω σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση σε σχέση με την γεωργία και τη δασοκομεία είναι σφαλμένη επιλογή. όπως είπε η κυρία η γεωργία είναι κομμάτι της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Και επίσης έχουμε δει ότι σε πολλά κράτη-μέλη όπου εφαρμόστηκαν ε, προγράμματα συντονισμένης δράσης περιβάλλον γεωργία, έχουν φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλω να ληφθεί υπόψη και να πούμε ότι οι προτάσεις πρασινίσματος που προβάλλονται τώρα εν ώψη της μεταρρυθμίσης στη γεωργική πολιτική είναι ευπρόσδεκτες ασφαλώς. Είναι σημαντικό όμως επίσης και να αναφέρουμε ότι τα μέτρα αυτά μπορεί για όλα εκείνα τα κράτη τα οποία ήταν στο παρελθόν διατεθειμένα και προέβησαν πράγματι σε μεγάλες προσπάθειες υπέρ της οικολογίας για το περιβάλλον δηλαδή είναι κακό μήνυμα. Ε, επίσης, στη γεωργία και το περιβάλλον ε, πολλούς άλλους τομείς που είναι σχετικοί και συνδεδεμένοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας για τον θα είναι υποχρεωτικές ή μη διατάξεις. Και επίσης πολλά είναι τα προβλήματα που σημειώνουμε σε σχέση με το σεβασμό των ε, διατάξεων και σε διεθνέ επίπεδο ακόμη, είναι λίγες οι ε, παραχωρήσεις των κρατών ε, σε διεθνέ επίπεδο, των τρίτων κρατών δηλαδή και οι προσπάθειές τους για τον περιορισμό παραδείγμα των εκπομπών θερμοκηπίου. Χρειάζεται λοιπόν μια γενικότερη συστράτευση για να βρεθεί, να δοθεί η σωστή και μεγάλη λύση. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαπραγματευόμαστε βεβαίως ε, σε σχέση με τρίτα κράτη. Ε, είναι πολύ μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος σε όλες μας τις διεθνείς συμφωνίες και νομίζω ότι πρέπει ακόμη περισσότερο να προβάλλουμε τη διάσταση περιβάλλον. Επίσης, η αναθεώρηση στρατηγικής για τη δεσοκομεία, για τα μάλλον σε συσχετισμό με, με τα περιβαλλοντικά προγράμματα έχει πολύ μεγάλη σημασία ώστε να μην ανατρέπονται οι στόχοι των περιβαλλοντικών προγραμμάτων από την πολιτική δασοκομεία. Πρέπει να, επιζη... Ε, να παρακολουθούνται οι παραλληλισμοί αυτοί και να αποτρέπονται αντίξω αποτελέσματα. Η καλλιέργεια της γης, η γεωργία εν είναι πολύ σημαντική και για την ε, παραγωγή ενδιαιτημάτων, χώρου διαβίωσης που προσφέρουν. Έτσι λοιπόν, χωρίς να περιορίζεται η παραγωγικότητα της γεωργίας, πρέπει να ε, κοιτάξουμε την διαχείριση των γεών, την αξιοποίηση, τις μεθόδους αξιοποίησης των γεών και πάνω απ' όλα ε, να ε, προσέξουμε όπου υπάρχει ζήτημα ε, περιορισμού των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, δηλαδή περιορισμού των φιλοξενούμενων σε ένα οικοσύστημα ή σε ένα ενδιαίτημα ειδών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ελίζαμπετ, Όσλιγκεν και μετά Μαγκίνες. Κύριος Χόισλιγκεν. Ναι, Πρόεδρε, ασφαλώς ε, κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ε, εδώ ότι οι σύγχρονες μορφές της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι πάντα κάτι το θετικό, οπότε εδώ βρίσκουν ε, ως αρνητική προοπτική. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι και κομμάτι της λύσης μπορεί να είναι η γεωργία, αλλά και κομμάτι του προβλήματος. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, γιατί θεωρώ ότι με την έκθεσή της σε μεγάλο βαθμό προσφέρει υλικό για σκέψη και μελέτη. Ιδιαίτερα στο θέμα της αγωγής πρωτεϊνών και τις συζητήσεις που γίνονται αλλά δεν ε, ολοκληρώνεται τελικά ποτέ το ζήτημα και δεν καταλήγουμε σε μια συμφωνία για το τι χρειαζόμαστε ως πρωτεΐνες στην Ευρώπη και σε ποιο βαθμό αρκεί η δική μας παραγωγή πρέπει να εισάγουμε από τρίτες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, εμεί υποστηρίζουμε τι θέσει τη εισηγήτρια. Ε, έχουμε θετικά βέβαια στοιχεία να προβάλλουμε σε σχέση με, τη γεωργία, με την δράση τη γεωργία, σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τα αρνητικά. Επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, διάρρηξη της τροφικής αλυσίδας, όπως το τελευταίο σκάνδαλο με ε, την παρουσία ε, κρέας αλόγου, κρέατος αλόγου σε συσκευασμένα τρόφιμα στην Ευρώπη. Και αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και να δούμε αν η νοοτροπία που έχουμε σε σχέση με τα τρόφιμα, την παραγωγή και διάθεση των τροφίμων είναι μια επιλογή σωστή και ορθολογική. Πάντως βλέπουμε ότι ο Γεωργός πιέζεται γιατί πρέπει να παράγει όλο και περισσότερο και θεωρώ βέβαια ότι δεν είναι σωστή η λύση αυτή γιατί πρέπει αντί για τις ε, βιοτεχνικές, ε, βιομηχανικού τύπου εντατικές παραγωγές να περάσουμε σε μια οικολογικά εντατική ε, γεωργία, δηλαδή με περισσότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα στη γεωργία. Από την άλλη, εάν διαπιστώνεται, όπως μας λέει και η συγκήτρια, ότι 50% των τροφίμων που παράγονται στην Ευρώπη δεν καταλήγουν στο πιάτο του καταναλωτή, τότε θα πει ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ λάθος και πρέπει να βρούμε λύσεις για να διαχειριστούμε καλύτερα αυτούς τους πόρους. Ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία των εδαφών που ακούστηκε νωρίτερα. Ασφαλώ έχει θέση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να πω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να συζητήσουν το θέμα τη προστασία των εδαφών ω ζήτημα αρμοδιότητα τη ευρωπαϊκή γεωργία και προσπαθούν να παρεμποδίσουν την περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση του θέματος αυτού ή την υποβολή προτάσεων. Πράγμα το οποίο είναι τελείω λάθο. Ε, με ένα κράτη όμω αν είναι το ζήτημα αυστηρά εθνικό και να μπορεί να περιοριστεί μέσα στα εθνικά σύνορα. Ενώ η καλύτερη λύση θα δοθεί μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Μαγκίνε και μετά Γιάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι συνδέεται με αυτή τη γνωμοδότηση για τη βιοοικονομία που θα αναλάβει η Επιτροπή μας και για να είμαστε συνεπείς θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. σχέση με τις τροπολογίες πιστεύω ότι όταν διαγράφουμε το intensive για τη γεωργία και γράφουμε βιώσιμες γεωργικές μεθόδους, εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για την παραγωγή ενέργειας και για τις μεταφορές δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αξιολογήσουμε το σύστημα είναι καλό ή κακό, γιατί πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε και οι διεργασίε ε, δεν είναι βιώσιμε. και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη διατύπωση ότι όλε οι σύγχρονε μέθοδοι έχουν καλά και κακά στοιχεία. Ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατύπωση. Για τα απόβλητα τροφίμων ε, συμφωνούμε όλοι ότι συνιστά αυτό το πρόβλημα και ο, ο Μάρτιν Χόσλινγκ είπε ότι 50% ε, των τροφίμων τα πετάμε στο σκουπιδοντενεκέ και λοιπόν ε, ε, ίσως επειδή είναι τόσο φτηνή, να τα τρόφιμα, τα πετάνε τόσο εύκολα οι άνθρωποι. Ε, σε σχέση τώρα με τις ε, τροφοδοτικές ε, αλυσίδες, Νομίζω ότι θα υπάρξει μία αντίδραση σε σχέση με το κρέας αλόγων. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η άποψή τους για να, συ... να ε, καταστεί πιο σύντομη η αλυσίδα, πιο μικρή η αλυσίδα και έτσι να καταστεί και πιο ασφαλής. Ε, στην ε, τροπολογία 25 μιλάμε ότι θα πρέπει να δώσουμε οικονομικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των αγροκτημάτων. Πολλά πράγματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στη Γεωργία απορρέουν από τις μεθόδους που εξυγχρονίστηκαν ναι μεν, όμως δεν αντιληφθήκαμε εμείς τις ε, επιπτώσεις ε, της εφαρμογής τους ε, και σε σχέση τώρα με την προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης βιωσιμότητας θα πρέπει οι γεωργοί να συνεργαστούν και με τους ερευνητές καθώς και με τους φορείς της αγοράς γιατί εκείνοι μπορούν να μας δώσουν τις σωστές απαντήσεις στα ερωτηματικά μας. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Κάτι άλλο σε σχέση με τις πληρωμές για τα δημόσια αγαθά. Τα τρόφιμα είναι δημόσια αγαθά. Ε, όταν ε, μιλάμε για την αγορά, δεν μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε μια σωστή τιμή για τα τρόφιμα αν δεν συνυπολογίσουμε και αυτό τον παράγοντα σε σχέση με τις άμεσες σχέσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές σε μέρος της τροπολογίας 7, ναι, θα ενθαρρύναμε κάτι τέτοιο, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και πιο ρεαλιστές. Ε, δηλαδή με ποιο τρόπο αγοράζουν ε, οι καταναλωτές τα τρόφιμα που για να λειτουργήσει εύρυθμα το σύστημα, όσοι έχουν άμεσες σχέσεις με τον παραγωγό, ε, είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που προμηθεύονται τα τρόφιμα σε υπεραγορές ε, και ε, σε διάφορα άλλη μέρη. Νομίζω ότι μέρος της λύσης για αυτά τα προβλήματα που εντοπίζουμε μέσα στην έκθεση εντοπίζεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και να προσαρμόσουμε τη διατύπωση. Σας ευχαριστούμε. Μαρίνο Πέτριγιαρ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την παρουσίαση Κάποιες παρατηρήσεις από πλευράς μου. Για να δώσω κάποιες ενδείξεις προς την τοποθέτησή μου. Εγώ θεωρώ ότι η γεωργία είναι κομμάτι του ε, της λύσης και όχι του προβλήματος ε, και χωρίς τη γεωργία δεν μπορούμε να βρούμε ε, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που έχω να επισημάνω. Πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Γιατί χωρίς ένα σύστημα γεωργικής παραγωγής δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης η ε, οικολογία. Και υπάρχει δυνατότητα με θελοντική συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, όπως άλλωστε αναπτύχθηκαν και στη Γερμανία, να βοηθήσουμε τον γεωργό να ε, συμβάλλει στην βελτίωση του περιβάλλοντος. Τώρα με το greening, ε, με το 7% και την αναλασσόμενη ε, υποβολή σε καθεστώς προστασίας κάποιων εκτάσεων κάθε φορά, πιστεύω ότι θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα ουσιαστικά, γιατί η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να αφορά ολόκληρη την καλλιεργούμενη έκταση, την υποεκμετάλλευση έκταση και όχι ένα μόνο κομμάτι της. Πάντως πρέπει να πω ότι οι εισαγωγές προϊόντων που δεν προέρχονται από αηφόρο παραγωγή και μάλιστα του αντίον ξέρουμε ότι μερικές φορές είναι τόσο δατική η καλλιέργεια ή παραγωγή που ε, καταστρέφει το περιβάλλον ε, στην περιοχή από την οποία προέρχονται τα προϊόντα. Εμείς όμως δεν έχουμε το θάρρος να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να πούμε ότι επιβάλλουμε τις ε, προϋποθέσεις για την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος που ισχύουν και στα δικά μας προϊόντα σε όσα είναι ε, εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Και επίσης ως προς τις ε, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην πέφτουμε στην παγίδα να χωρίζουμε την γεωργία σε καλή και κακή, δηλαδή άλλοι να είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά στο περιβάλλον και κάποιοι άλλοι καταδικάζονται γιατί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Πρέπει να δούμε οι νέες τεχνολογίες που θα προτείνονται να φέρουν πραγματικά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ανάλογα με το μέγεθος, της εκτάσεις δηλαδή, ε, και ως προς τα αποτελέσματα και ως προς, το επιδιωκόμενο, ως προς την επιδιωκόμενη τελικά προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά θα θετυπώσουμε τις απαραίτητες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Δεν είστε άλλο το λόγο από τους συναδέλφους και γι' αυτό παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ε, κύριο Βετόρη από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για να δώσω το λόγο στη συνέχεια στην κυρία Σάρβο. Κύριε Βετόρη, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President, for... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. Και ευχαριστώ και την ε, κυρία Σάρμπου για το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ο στόχος ε, της Επιτροπής με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον ήταν να θέσει ένα πλαίσιο για να εκπονηθούν πολιτικές δείχνοντας ε, με ποιο τρόπο οι διάφορες πτυχές των επιμέρους πολιτικών είναι αλληλένδετες, ε, συμβάλλοντας ε, έτσι όχι μόνο σε ένα καλύτερο ε, περιβάλλον αλλά και στην ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Δείχνουμε ότι η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πορών συνδέεται με την προστασία της βιοπικιλότητας και του περιβάλλοντος αναβαθμίζοντας την ανθρώπινη υγεία και υποβαθμίζοντας τους χημικούς κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα οικοσυστήματα σε τις προτεραιότητες μέχρι το 2020 θα επιτευχθούν από τα κράτη-μέλη, από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως ε, μην ξεχνούμε ότι η γεωργοί είναι πολύ σημαντικοί ε, παίκτες ε, στην προσπάθεια που κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρχίζουμε κάνοντας την ανάλυση επί τη βάση της έκθεσης Τη ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ε, ε, τονίζοντας ποια είναι τα υφιστάμενα κενά κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τις προτεραιότητες για το 2020, όπως σας έλεγα, κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογιστεί. Για να επιτύχουμε τις προτεραιότητες, αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερο από έναν μακρύ κατάλογο προτάσεων ή λεπτομερών πρωτοβουλίων πληροφοριών εκτιμούμε το ότι αναφέρεστε στην έκθεσή σας στα απόβλητα τροφίμων. Είναι και για μας πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και επεξεργαζόμαστε τώρα μια ανακοίνωση που θα εκδοθεί τους προσεχείς μήνες για τα απόβλητα τροφίμων, κάνοντας μια αναφορά φυσικά στην ε, βιώσιμη γεωργία. Το έδαφος. Το έδαφος είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η ποιότητα του εδάφους έχει κέρια σημασία για την αποθήκευση του άνθρακα, για την καλλιέργεια, για την προσαρμογή κλιματικές ε, αλλαγές, ε, για την, ε, τον καθαρισμό των λιμάτων και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικά στοιχεία λοιπόν για τη μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Ως προς τροπολογίες, ε, εν γέννη μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Στην τροπολογία 3 θα προτιμούσαμε να αναφερθούμε σε όχι να αναφερόμαστε στη γονιμότητα του εδάφους αλλά στα οργανικά στοιχεία που έχει το έδαφος διότι όταν μιλάμε για την γονιμότητα υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν σε αυξημένη ρήπανση και όχι σε αυξημένη βιωσιμότητα. Τροπολογία 5. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η καινοτομία για την βιωσιμότητα της μελλοντική ε, γεωργικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως θα πρέπει να μην περιοριστούμε στην ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αλλά να αναφερθούμε και σε σημεία όπως παραδείγματος χάρη ο γεωργικός εξοπλισμός. Τροπολογία 7 εκεί βλέπουμε την άμεση σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή και ότι μπορεί αυτό να συμβάλλει σε πιο βιώσιμη κατανάλωση ε, των τροφίμων και όπως σωστά είπαν κάποια μέλη της Επιτροπής σας, αυτή δεν θα είναι και η μοναδική ευκαιρία που θα έχουμε για να επιτύχουμε τον εν λόγω στόχο. Τέλος, ως προς τα απόβλητα τροφίμων στην τροπολογία που προτείνεται η καταληκτική ημερομηνία είναι το 2005 για να μειώσουμε κατά το ίμιση τα απόβλητα τροφίμων στην Ένωση. Πιστεύω ότι για να είμαστε συνεπείς με την καταληκτική ημερομηνία του Κοινοβουλίου που συμπεριλήθηκε στην έκθεση για ε, τα απόβλητα τροφίμου του Σαλβατόρα Καρόνα ε, το 2011. Θα πρέπει να θέσουμε τον ίδιο στόχο. Το 2025 θα πρέπει να είναι η καταληκτική ημερομηνία και όχι το 2030 διορθώνει το ο όπως αναφέρεται μέσα στην τροπολογία. Ε, ως προς τις επιδοτήσεις, ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις προτινόμενες από, την εισηγήτρια αλλαγέ, ε, διότι αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρή περιστολή των επιδοτήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγγραφούν σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο οι επιδοτήσεις. Παραδείγματος χάρη, επιδοτήσεις ε, για εταιρικά οχήματα και άλλες τέτοιες κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη πρωτοβουλίες ε, ε, για τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να συμπεριληφθούν. Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες εν που αναφέρονται μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, προσβλέπουμε στην ε, συνέχεια της διαδικασίας και στην μελλοντική ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Βετόρη. Η συγγήτριά μας έχει τώρα το λόγο για την καταληκτική της παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστώ του συναδέλφου για τι πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει του και τα σχόλια. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να είναι αρνητική η στάση μας ή ο τόνος στο κείμενο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι τροπολογίες, να κάνουν τις προτάσεις τους οι συνάδελφοι, να συμμετάσχουν. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι πολύ σαφής η στόχη μας να μιλάμε λιγότερο και να κάνουμε περισσότερο. Χαίρομαι που δέχεσαι την πρότασή μου για τον ρόλο ε, στην προσφυγή του περιβάλλοντος και της δαξοκομείας, όπως και της γεωργίας. Και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να περιοριστούν ε, τα απόβλητα από τρόφιμα. Γι' αυτό ιδιαίτερα είμαι υπέρ της ε, πιο μικρής σε απόσταση αλυσίδα τροφίμων, δηλαδή κατανάλωση των προϊόντων στην τοπική τους αγορά. Γιατί μεγάλο κομμάτι από αυτό που χάνεται από τρόφιμα έχει να κάνει με τις μεγάλες αποστάσεις από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ βέβαια να κάνω σχόλια σε όσα είπαν οι συνάδελφοι, τα σημείωσα όμως όλα. Είμαι στη θέση τη συζήτηση και ελπίζω ότι η πρόταση που θα καταθέσω εν τέλει να είναι ικανοποιητική για όλου του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Και προχωρούμε έτσι στο επόμενο θέμα τη σημερινή διάταξη, το υπαριθμό 6. Ετήσια έκθεση για το 2011 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Βοσεβόσκη μαζί με την ετήσια έκθεση ή που αφορά καλύτερα την ετήσια έκθεση του 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση. Προτείνεται η διαπίστωση ότι έχουν μειωθεί στο μισό περίπου οι παρατυπίες που καταγράφονται και τα τόσο καταβληθέντα ποσά για το 2011 για όλους τους τομείς 1.230 παρατυπίες καταγράφονται ως ε, προϊόν απάτης. 35% ε, λιγότερο από το 2015 δηλαδή, ε, από το 2010 συγγνώμη. Θα παρακαλέσω τον εισηγητή να λάβει το λόγο, τον συντάκτη της νομοδότησης, για να αρχίσει μετά η συζήτηση. Ευχαριστώ. με την ε, ε, ιδιότητα του εισηγητή ασχολήθηκα με ένα τμήμα μόνο αυτή τη έκθεση που σχετίζεται με την σφαλμένη χρήση των πόρων στον τομέα της γεωργίας, διότι βλέπουμε στην έκθεση το 2011 από όλες τις παρατυπίες 2.395 το αριθμό η 139 είναι ε, καταχρήσεις σε σχέση με την κατάσταση το 2010 παρατηρήθηκε μείωση των παρατυπιών ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις αυξήθηκαν 77 εκατομμύρια ευρώ το 2011. Στην έκθεσή μου επικεντρώνομαι σε κάποια ιδιαίτερα ε, σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως οι πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει τα κράτη-μέλη ενδέχεται να μην είναι πλήρως αξιόπιστες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει δε ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι παρατυπίες είναι ελάχιστες. Ίσως αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το κράτος μέλος ε, ε, δεν ε, ταξινομούνται με τον ίδιο τρόπο οι καταγγελίες ως παρατυπίες δηλαδή ως κάτι άλλο. Ε, άρα ε, το σύστημα υποβολής αναφορών για τα στοιχεία των ε, κρατών μελών θα πρέπει να αναθεωρηθεί ούτως ώστε να έχουμε ομοιόμορφα στοιχεία από πλευράς των κρατών μελών σε σχέση με την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών. Για να αποτραπούν μελλοντικέ παρατυπίες και ε, καταχρήσεις ε, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε μόνο στατιστικά εργαλεία και στατιστικά δεδομένα. Θα ε, έπρεπε να εφεύρουμε νέους μηχανισμούς, μια νέα υποδομή, ούτως ώστε να επεξεργαζόμαστε τις σοβαρότερες παρατυπίες κατά προτεραιότητα. Βασίζουμε επίση τα συμπεράσματά μα, ξαναλέω, αποκλειστικά και μόνο σε στατιστικά στοιχεία, κάτι που να ο Γιούλιαν Τούβιν, ένας Πολωνός ποιητής, είπε ότι υπάρχουν τρία είδη ψεμάτων. Ε, το κοινό ψέμα, το ε, ψέμα όταν κάποιος έχει ορκιστεί και το, η τρίτη κατηγορία, λέω εγώ, θα έπρεπε να είναι το στατιστικό ψέμα. Η παραποίηση δηλαδή των στατιστικών στοιχείων, διότι έτσι παραποιείται η εικόνα που παρουσιάζεται για την αποτίμηση της κατάστασης δεν θα έπρεπε η Επιτροπή να βασίζεται ε, μόνο σε στατιστικά στοιχεία αλλά και σε ποιοτικά. Ο Γάλλος δεν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης και δεν θα γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποια είναι τα προβλήματα. Ε, γι' αυτό προτείνω να κάνουμε μια υπέρβαση σε σχέση με την αποκλειστική χρήση των στατιστικών στοιχείων. Αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο της έκθεσής μου. Άλλα σημεία κλειδί στην έκθεσή μου ε, σχετίζονται με την αξιοπιστία, Φερρυπίνε, των στατιστικών στοιχείων που ε, διαβάζουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι και αυτό δημιουργεί με λανθασμένη εικόνα. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα της στατιστικής ανάλυσης. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε περαιτέρω, ε, διότι είναι ανεπαρκές το σύστημα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο. Ο Γιάννη ζήτησε το λόγο. Μια στιγμή παρατήρηση εδώ. Ναι. Για το όσο υποσηγητής, ευχαριστώ. Καταρχά. και νομίζω ότι έθεσε το δάκτυλο από τον τύπο των ήλων ο εισηγητή. Έχει διατυπώσει σαφεί προτάσει που ήταν και τροσιώτε για μένα, διότι εάν δεν υπάρχει ένα ε, ενιαίο ορισμό στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι σημαίνει ουσιαστικά πάτη ή απόπειρα απάτης, πώς δηλαδή θα καταγραφεί η απατηλή συμπεριφορά, τότε οποιαδήποτε στατιστική δεν έχει καμιά αξία. Και έτσι αρχίζει μια ένα αγώνα τρόμου προ τα κάτω των κρατών μελών, δηλαδή να δηλώσουν στο δυνατόν λιγότερε περιπτώσει απάτη. Θέλοντα ότι θα παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα. Για μένα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το κομμάτι εκείνο στο οποίο γίνεται λόγος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου αυτή καλείται να καταγράφεται η απάτη με ακριβείς, τρόπο, με ακριβείς τρόπους και με ακριβείς ορισμούς. για να μην έχουμε τελικά το φαινόμενο της ρουλέτας, άλλος να δηλώνει, άλλος να μην δηλώνει και τελικά αυτός που έχει δηλώνει την πρώτη απάτη, να φαίνεται ότι την πάτησε τελικά. Γιατί εκτίθεται. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο να είναι καθαρά στις ε, δηλώσεις του, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζει όταν δηλώνεται μια ε, παραβίαση, μια ε, πατελή περιφορά, Αυτή θα ισχύει με τους ίδιους όρους για όλους. Ξέρετε ότι συνήθω λέγεται ότι η μόνη στατιστική μπορεί κανεί να, να εμπιστευτεί είναι αυτή την οποία έχει ο ίδιο παραποιήσει. Ελπίζω να μην ισχύσει αυτό στην περίπτωση των στατιστικών για, τις, ε, για τα θέματα του προπολογισμού. Χάρη και στον ε, εισηγητή, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλά στοιχεία. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί, κυρία Μαγκίνε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Με ανησυχεί αυτή η παράγραφος 4. Ε, ο εισηγητής λέει ότι οι περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως απάτη σε, κάποια, σε, σε κάποια κράτη-μέλη θεωρούνται νομότυπες σε άλλα. Έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Να ρωτιέμαι Έχω την εντύπωση ότι είναι μάλλον ανέφικτο αυτό που ισχυρίζεστε και άρα θα χρειαστούμε μία έκθεση για αυτή την παράγραφο αν ισχύουν αυτά που ε, προτάσετε εδώ. Έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη. Αν όντως αληθεύουν, χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Ε, δεν μπορεί ε, σε ένα κράτος μέρος να θεωρείται κάτι έκνομο και σε άλλη σύνομο. Ευχαριστώ. Σημαντικό θέμα. Καπούλα Σάντος πρώτα. Ευχαριστώ. Ε, συγχαίρω και εγώ τον ε, εισηγητή γιατί είναι πολύ κέρια τα ζητήματα που γύρει και θα ήθελα να ε, προσθέσω στον κύριο, και αναφέρομαι στον κύριο Γέρμη έναν άλλο ορισμό των στατιστικών στοιχείων. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και μελετούσα τη στατιστική, ο κύριος Κίτλη είχε προτείνει ένα νέο ορισμό η τέχνη του να ψεύδεται κανείς με ακρίβεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε, ε, ε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με τη στατιστική ανάλυση. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε για ποιο λόγο θέλουμε ε, να απλουστευτεί η κυνηγεωρική πολιτική. Όσο πιο περίπλοκη είναι η γραφειοκρατία, τόσο πιο δύσκολα εντοπίζουμε τις παρατυπίες. Όπως είπαν οι συνάδελφοι και κυρία Μαγκίνες που μίλησα τώρα τελευταία, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, είναι σημαντικό αυτό που ισχυρίζει ο εισηγητή, ότι υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα ήθελε ο εισηγητή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσουν κάποιε επιπρόσθετε πληροφορίε σε σχέση με ε, αυτά τα διαφορετικά κριτήρια που φαίνεται να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον έλεγχο και την πάταξη τη απάτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίντρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή πραγματικά για τη δουλειά του. Ο κύριος Βοητσεχόφης έκανε πολύ καλή δουλειά. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνεκτική εικόνα της κατάστασης σε όλη την Ένωση. Αναγνωρίζω, όπως και άλλοι ομίλητες, τον ορισμό του για την στατιστική. Τα τρία επίπεδα στην Βρετανία ε, έχουν την εξής ε, ιεράρχηση. Ψεύδι, μεγάλα ψεύδι και στατιστικές. Άρα βλέπετε ότι όλη την ίδια ανάγνωση έχουμε. Επίσης, ήμουν στην Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματο και την οργανωμένη εγκληματικότητα και ως κοινοβούλιο μπαίνουμε όλο και περισσότερο στο να καταλαβαίνουμε καλά το οργανωμένο έγκλημα διευρωπαϊκά. Η κοινή γεωργική πολιτική προφανώς ε, αντλεί ένα τεράστιο ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης. Είναι σημαντικός τομέας για να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Επίσης, να υποστηρίξω τους προηγούμενους ομιλητές για να γίνει πιο συνεκτική και απλούστερη παρακολούθηση, πρέπει να υπάρχει μια απλοποιημένη κοινή γεωργική πολιτική με απλούς κανόνες, ούτως ώστε να τηρούνται σε όλη την Ένωση με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δεν το κάνουμε και αυτό οδηγεί συχνά σε αποσυντονισμό του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζουν τις αιτήκες τα κράτη-μέλη. Καλό λοιπόν να, υπήρχε, να υπάρχει μια μεγαλύτερη απλοποίηση για να υπάρχει και συνεκτικότητα σε όλη την έννοιση. Ε, ευχαριστώ πάντως ξανά τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Ωραιότατα. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Βάντερ Φέλστ από την Όλαφ και Μπάντερ από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Ποιος θέλει το λόγο από εσά. Κομισιόν. Παρακαλώ. Κάνουν διαβουλεύσεις. Ε, good afternoon. Thank you for... Ε, Καλησπέρα και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Κάποιες παρατηρήσεις από πλευράς μας. Να σας πω και ποιος είμαι πρώτα. Φέλς λέγομαι. Είμαι υπεύθυνο για την στατιστική ανάλυση, τη σύνταξη της στατιστικής ανάλυσης του τμήματος Γεωργίας. Επίσης ανήκω στη Γενική Διεύθυνση Ανάλυσης ε, της ΟΛΟΦ και είμαι υπεύθυνο για στατιστικά. Στατιστικά στοιχεία που ορισμένοι περιέγραψαν εδώ ως ε, την ανώτερη βαθμίδα του ψεύδους. Άρα δεν είμαι μεγάλος ψεύτης, κάνω στατιστικά. Για να απαντήσω στα σχόλια. Πρώτον, ζητούμε από τα κάτι μέλη να ταξινομούν τις ατασταλίες. Εμείς το βλέπουμε ως εξής. Έχουμε ατασταλίες και μέσα στο σύνολο υπάρχει το υποσύνολο υποψία απάτης. Η υποψία απάτης περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου υπάρχει ε, πρόθεση ε, διάπραξης ατασταλίας. Υπάρχει άλλο υποσύνολο μέσα στην ομάδα. Η υποψία απάτης, δεδομένη, καθιερωμένη απάτη, όταν υπάρχει δικαστική απόφαση, άρα έχουμε τρία επίπεδα. Η υποψία απάτης, με πρόθεση και απάτη όταν υπάρχει πια δικαστική απόφαση. Συζητήσαμε με τα κρατημέλη σε, διάφορα, σε διάφορες συναντήσεις, μεταξύ των οποίων τις αμοιβέ συνδρομής της και ατασταλής στα γεωργικά προϊόντα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα τι συζητάμε. Ένα θέμα που περιλαμβάνεται στο σημείο 4 της έκθεσης ζητήθηκαν ε, παραδείγματα. Και μπορώ να σας πω ότι συζητήσαμε στην τελευταία συνάντηση της αμοιβαία συνδρομής που έχει το 1848 ακρόνιμο βάση του κανονισμού πάνω στον οποίο στηρίζεται είναι ξεκάθαρη. Η επιδότηση των γεωργικών προϊόντων στηρίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί εφαρμογή των κανόνων που θέτει η Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την ίδια νομοθεσία για να αναφέρουν τις ατασταλίες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν στο α κράτος μέλος να θεωρείται νόμιμο νόμιμη μία πράξη, μία συμπεριφορά και σε, και σε άλλο κράτος να θεωρείται ατασταλία. Και αν πραγματικά σημαίνει κάτι τέτοιο θα με εξέπλητε. Τα κράτη-μέλη πάντως διστάζουν να αναφέρουν ή να ταξινομούν ατασταλία ως, ως υποψία απάτης λόγω του ότι φοβούνται μήπως ε, δυσχεράνουν μια υποεξέλιξη ανάκριση ή έρευνα δικαστική έρευνα. Επίσης να αναφέρουμε ότι το στατιστικό παράτημα είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της δουλειά που κάνουμε. Δεν παρέχουμε δηλαδή στατιστικές, κάνουμε και άλλες δουλειές. Δυστυχώς η έκθεση πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα η προθεσμία που έχουν τα κρατημέλη για να υποβάλουν ε, τις ατασφαλίες είναι 28 Φεβρουαρίου και μετά έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να συμπεριλάβουμε τα πάντα στην έκθεση. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν κάνουμε και άλλες αναλύσεις, περαιτέρω αναλύσεις, ίσα ίσα. Αυτό που βλέπετε απλά είναι κάτι πολύ πιο ε, βασικό. Λοιπόν, ναι, κάνουμε πολλά πράγματα πέραν των ε, στατιστικών σε αναλύσει, αλλά αυτά δεν εμφανίζονται στην έκθεση. Γιατί δεν είναι ο σωστός χώρος, το σωστό πλαίσιο. also good uh, to mention that uh, the impact of the two cases mentioned in point one. να αναφέρουμε και ότι ο αντίκτυπος των δύο εκθέσεων που αναφέρθηκαν στο σημείο 1 περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις όπου ξεκίνησε η ανάκτηση του 2003 όταν έγινε αναφορά των ε, περιπτώσεων αυτών το 2011 γιατί σας είπα ότι κράτησαν ε, οι έρευνες τόσα χρόνια και δεν ήθελαν να πλήξουν τις ε, έρευνες. Οι δύο αυτές ε, περιπτώσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό νούμερο για το 11, οπότε καλό ήταν να τις αφαιρέσουμε για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Κάτι άλλο. Η έκθεση αφορά, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν Γαλλία και Ολλανδία. Και στην Ολλανδία έγινε αναφορά από, από την Ολλανδία έγινε αναφορά το 2011, οπότε και πάλι έχεις μία απόκληση που προκύπτει από την επανεμφάνιση της ίδιας υπόθεση. Μήπως θες να πεις κάτι άλλο εσύ συνάδελφε. Ευχαριστώ. Και όλα λέγουμε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Εμείς κάνουμε παρακολούθηση, οικονομική παρακολούθηση και σωστή ανάκτηση από πλευράς εθνικών αρχών των ατασταλιών. Χωρίς να μπω στη διάκριση διαπιστωμένη απάτη, υποψία απάτης ή ατασταλία, εμείς θέλουμε να ε, εμείς απάτηση, η ανάκτηση των κονδυλίων γίνεται με σωστό τρόπο από τους οργανισμούς πληρωμής και από τις εθνικές αρχές. Όπως είπατε Πρόεδρε, η ανάκτηση από τους δικαιούχους, ε, σε ό,τι αφορά την ανάκτηση από τους δικαιούχους βελτιώνεται η κατάσταση υπάρχει καταμερισμένη διαχείριση της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά η ανάκτηση εξαρτάται, συνεχίζει να εξαρτάται εμπολής από την εθνική νομοθεσία και από τις εθνικές ε, ρυθμίσεις ε, τόσο δικαστικού χαρακτήρα όσο και αποζημίωσης. Για την περίοδο 14-20 η Επιτροπή προτείνει να προχωρήσουμε παραπέρα διευκρινίζοντας ορισμένους κανόνες ότι αφορά την πληρωμή, την ανάκτηση αδικαιολογήτως καταφληθέντων και την αλλαγή του υφιστάμενου κανόνα 50-50 που είναι ότι το 50% των κονδυλίων που τα κράτη δεν ζητούν πίσω ε, μπαίνει στον εθνικό ή μάλλον αφαιρείται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Εμείς θέλουμε όλο το ποσό που δεν ανακτάται από το κράτος μέλος να χρεώνεται στο κράτος, στον προϋπολογισμό του κράτους μέλος, τόσο ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τον προϋπολογισμό της Ένωσης και να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, ούτω ώστε να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν οι εθνικές αρχές την διαδικασία ανάκτησης των ε, αχρεωστήτων καταπληθέντων. Αυτά. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβαση των εκπροσώπων της Επιτροπής και της Όλαφ. Δίνω τώρα ξανά το λόγο στον συνάδελφο Βαϊσεκόφσκι και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Γιάννους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις δηλώσεις και τις προτάσεις τους σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης. Ε, για την κυρία Μαγκίνες θα ήθελα να απαντήσω ε, για, σε αυτό που μου είπε για την παράγραφο 4 ότι δηλαδή ενδέχεται να διαφέρουν τα κριτήρια που εφαρμόζονται για ταξινόμηση των περιπτώσεων των παρατυπιών. Δεν έχω εις βάθος γνώσης για το ζήτημα αυτό. Βασίστηκα όμως ε, στη δήλωσή της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εκεί ο εισηγητής ε, στην εχνομοδότηση του εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξημένο αριθμό παρατυπιών ε, στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σταριστικός πώς φαίνεται ότι δεν είναι ε, ξεκάθαρη η κατάσταση διότι ε, είναι δυσανάλογος ο αριθμός των παρατυπιών σε σχέση με το μέγεθος ε, των αγροκτημάτων ή τον αριθμό των παραγωγών σε κάποιες χώρες. Δεν έχουν δεν έχουν ε, αναφερθεί συγκεκριμένα κράτη-μέλη μέσα στην έκθεση της ε, Επιτροπής Ελέγχου των ε, Προϋπολογισμών. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό το σημείο και να εξετάσουμε εντελεχέστερα τον τρόπο ταξινόμησης των παρατυπιών. Από τη δικιά μου χώρα έχω κάποια εμπειρία και σας διαβεβαιώ ότι οι πολωνικές ε, αρχές ε, εμπλέκονται ενεργά στη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. 8.000 ε, περιπτώσεις έχουν διαβιβαστεί σε αρμόδιες αρχές και ελάχιστες μόνο οδήγησαν σε βεβαιωμένη απάτη. συντριπτική πλειοψηφία ε, σχετιζόταν με ε, περιπτώσεις όπου οι γεωργοί βασίζουν τις αξιώσεις τους ε, σε παροχημένα γεωφυσικά δεδομένα και οι σύγχρονοι χάρτες, δορυφορικοί χάρτες δεν ταιριάζουν με τα ιστορικά δεδομένα. Δεν πρόκειται δηλαδή για θελημένη απάτη. Ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα ίσως έδειξε υπερβολικό ζήλο για τη δίωξη των παρατυπιών και δημιουργήθηκε έτσι αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν σε άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχες εμπειρίες. Πιστεύω πάντως σε κάθε περίπτωση πως ε, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να παταχθεί η απάτη αν γίνεται ηθελημένα. Όσοι τώρα ε, ε έχουν παρατυπήσει ε, λόγω ανθρωπίνου λάθους ή ε, επειδή έχει διαπραχθεί κάποιο λάθος στις δηλώσεις τους θα έπρεπε να έχουν διαφορετική μεταχείρισης. Πιστεύω πάντως ότι στο μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει ε, αυτό το σημείο, διότι ε, όντως ε, μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και όντω μπορεί τα στατιστικά στοιχεία να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος κύριε Βοσικιώσκη και περνάμε στο σημείο 7.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 Ευχαριστώ και καλό απόγευμα σε όλους. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα καταδεικνύει πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα που πραγματευόμαστε. Είναι ξεκάθαρο. Εξ αρχή θα έπρεπε ίσω να ξεκαθαρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα βιώσιμα βιοκαύσιμα μπορούν να μειώσουν σε εκπομπέ αερίων θερμοκηπίων, μπορούν να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και να δημιουργήσουν βιωσιμότητα στον τομέα των μεταφορών. Ε, αυτές είναι, αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιοκαυσίμων και πρέπει να τα διασφαλίσουμε. Τι άλλαξε όμως ε, και εξάλλου κάποια μέλη της Επιτροπής το ανέφεραν αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή άλλαξε ρότα για τα καβιοκαύσιμα. Τι άλλαξε λοιπόν. Ε, γνωρίζουμε περισσότερα σήμερα σε σχέση με το 2008-2009 όταν διαπραγματευόμασταν για αυτήν την οδηγία. Ξέρουμε ότι αυτά τα έμεσα αποτελέσματα μπορούν να είναι αρκετά σημαντικά και ξέρουμε ότι συνδέονται με κάποια είδη βιοκαυσίμων, κυρίως της ε, πρώτης γενναίας που βασίζονται σε καλλιέργειες ε, πρέπει να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Ο δάλος θα, τα βιοκάσιμα θα χάσουν κάθε αξιοπιστία στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, θα, βρεθούν, θα είναι πολύ άσχημη η κατάσταση για τα βιοκάψιμα. Εμείς προτείνουμε μια σωστή απάντηση για τις προκλήσεις των βιοκαυσίμων σήμερα. Θέλουμε να περάσουμε ε, ένα ηχηρό μήνυμα στους γεωργούς τη βιομηχανία και σε όσους αναπτύσσουν νέες τεχνολογικές μεθόδους. Τα μελλοντικά βιοκαύσιμα θα διαφέρουν από τα σημερινά, διότι δεν θα βασίζονται σε καλλιέργειες, θα βασίζονται σε πρώτες ύλες που δεν, δεν έχουν έμεσες επιπτώσεις ε, όπως ε, αυτό που συμβαίνει ε, στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Υπάρχει εδώ και, και καιρό η πρόταση που κάναμε και αυτό πάλι δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Πάντως κατά τη γνώμη μας ε, εξισορροπούνται χάρη σε αυτή την πρόταση τα διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν στον τομέα των βιοκαυσίμων από πλευρά όλων των φορέων δηλαδή και των εμπλεκομένων φορέων. Ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάχνουμε οικονομικά μοντέλα. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε αν ευσταθούν αυτά που ισχυριζόμαστε διότι αυτό αιτιολογείται από την έλλειψη επιστημονικών στοιχείων ε, στον τομέα. Πάντως εμείς βασιζόμαστε στα ε, καλύτερα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Ας μπω σε κάποιες λεπτομέρειες για την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, προτείνουμε να μειώσουμε τα κίνητρα για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Δεν προτείνουμε να μειώσουμε ούτε την παραγωγή αλλά ούτε και την κατανάλωση αυτών, μόνο τα οικονομικά κίνητρα θα περικόψουμε περιορίζοντας τη... το βαθμό χρήσης των ε, βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς για να επιτευχθεί ο στόχος 10% που αναφέρεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια νέα κίνητρα για τα ε, για τον τριπλό και τετραπλό μέθοδο υπολογισμού και τα νέα βιοκάψιμα προσδιορίζουμε το τι θα συγκαταλεχθεί σε αυτές τις κατηγορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία που της έχει δώσει η ίδια βιομηχανία σε σχέση με το τι συνιστά απόβλητο, η κατάλοιπο και το καθεξής. Προσπαθούμε να κάνουμε μία πρόταση για να διαφυλαχθούν και οι επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει, διότι αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα σε διάφορες παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα είναι ότι προφανώς η βιομηχανία, η γεωργία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βασίστηκαν ε, στα συμπεφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πριν από λίγο καιρό ε, για τις επενδύσεις που θα γινόντουσαν και άρα πρέπει να τις διασφαλίσουμε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι χάνονται αυτές οι επενδύσεις τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς είναι, έχουν φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο 5%. Λοιπόν, θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε πιο... Ε, πιο εξελιγμένα ε, βιοκαύσιμα ε, και να εφαρμοστούν τα στοιχεία iLook. Οι παράγοντες iLook θα πρέπει δεν να προσμετρούνται με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Δεν είναι νομοτεχνικός ο στόχος. Ο στόχος είναι να επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον ε, κλάδο, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές τους επιπτώσεις ή οι εκτιμούμενες πραγματικές επιπτώσεις τους σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτά είναι σε πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, τα θέτει αυτές τις προτάσεις στο νέο πακέτο θα θέλαμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να βρούμε μια ε, ικανοποιητική λύση. Ξέρουμε πόσο ακαθόδες είναι το ζήτημα και πόσο ε, δύσκολο θα είναι να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στα διακριτά συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων ε, φορέων, αλλά είμαστε σίγουροι ότι σε στενή συνεργασία με τον κύριο Γκλάτ Φέρντερ και με τα υπόλοιπα μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής Γεωργίας θα καταφέρουμε τελικά να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα ακούσουμε ακούσουμε τον κύριο Κλατφέλντερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητέ για τη συνεισφορά τους και τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Έδωσαν μια ακριβέστατη παρουσίαση των θέσεών τους. Θέλω να λάβουμε υπόψη, θέλω να λάβω υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις όταν προχωρήσω περαιτέρω στο σχέδιο, στην επεξεργασία του ε, δύο εκθέσεις και θα το συντονίσω με όλους τους συναδελφούς όσο περισσότερο μπορώ. Πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν πιστεύει ότι είναι αξιόπιστες αυτές οι μέθοδοι υπολογισμού. Υπάρχει λοιπόν ευρεία συμφωνία ως προς το μη αξιόπιστο των υπολογισμών. Αλλά αυτό είναι βασικό θέμα που αντικατοπτρίζεται σε οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω δραστηριότητά μας. Κάθε μέτρο που υιοθετηθεί βάσει αυτών των υπολογισμών πρέπει να προϋποθέτει ότι θα γίνει συζήτηση των μέτρων αυτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αν εμείς έχουμε επιφυλάξεις για τους υπολογισμούς αυτούς, θεωρούμε δηλαδή ότι είναι αναξιόπιστοι κάθε μέτρο που στηρίζεται σε αυτό θα αποτύχει. Και εάν ένα μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει στο διεθνές εμπόριο, είναι προφανές ότι δεν αξίζει να το ε, δοκιμάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σενάριο λοιπόν θα πρέπει να το αποκλείσουμε για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα την γκράμβη και γενικότερα τους ελαιούχους σπόρους δεν είναι πρωτεϊνούχα φυτά. Τα υπολείμματα των συγκομιδών αυτών περιλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό πρωτεΐνης. Το ίδιο ισχύει και για το στάρι. 23-24% του σταριού είναι πρωτεΐνη. Αν αφαιρέσουμε το άμυλο, και αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, σαν πείραμα. Έπρεπε να αφαιρέσουμε το άμυλο από τα... στο στάρι και το υπόλοιπο ήταν, ήταν πρωτεΐνη. Έτσι δημιουργούμε και ποιοτικό αλεύρι εν τέλει. Οι ελαιούχοι σπόροι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα πρωτεΐνης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, αποτελεσματικά ως ε, χορτονομή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια τη ενέργεια που είναι θέμα που δεν είναι δικό μα, δεν πρέπει να αγνοηθεί. Είναι μια παράμετρο που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η Ευρώπη έχει πλεόνασμα πετρελαίου που πωλείται σε, σε χαμηλή τιμή στη διεθνή αγορά ενώ έχουμε έλλειμμα σε δίζελ. Η παραγωγή λοιπόν βιοδιζελ θα ήταν χρήσιμη από ενεργειακής απόψεως λοιπόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να είμαστε τρωτοί αν ε, δώσουμε έμφαση στην παραγωγή βιοντίζελ μέσω της διαδικασίας αλκοόλης. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι η απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να αναθεωρείται. Υπάρχει κάποιο χρονικό φυσικό σημείο το 2020 που ήταν η τελική ημερομηνία της αρχικής πρότασης. Η φυσική ημερομηνία μιας τέτοιας αναθεώρησης και αποψή μου μπορεί να είναι μόνο το 2020. Κάτι που επίσης θυμάμαι σαφώς είναι το εξής. Η Επιτροπή λέει ότι η πρόταση είναι ισορροπημένη και ότι έλαβε υπόψη κάθε διάσταση του θέματος. Αλλά πριν από 6-7 χρόνια ερχόταν η Επιτροπή και έλεγε τα ίδια πράγματα. Έλεγε ότι οι ανησυχίε για την εκπομπή του δημοσίου του, του ανθρώπου για την ασφάλεια των τροφίνων είχαν ληφθεί υπόψη. Και εγώ τότε ήμουνα κάποιο από αυτού του άπιστου θωμάδε. Η Επιτροπή μα έλεγε όχι, δεν είναι έτσι και τα έλεγε με την ίδια υπεροψία και ε, αιμονή όπως και τώρα. Ελπίζω ότι θα εξασφαλίσει μια σταθερότητα γιατί αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα για τους επενδυτές θα τους πείσουμε να επενδύσουν σε βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Παίζουμε με την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ. Ωραία συνάδελφοι. Τελειώσαμε νομίζω, δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Τελευταίο σημείο στη ημερησία διάταξη. Παρουσίαση από πλευρά Επιτροπή τη κατάσταση των εισαγωγών εσπεριδοειδών από την Κίνα. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στις 22 Μαρτιού το Δικαστήριο της Ένωσης ακύρωσε τον κανονισμό 1355 του 2008 που επιβάλλει οριστικό δασμό αντι-dumping και, και προσωρινούς ε, ε, δασμούς εισαγωγής σε ορισμένα προϊόντα εσπεριδοειδών είτε ε, φνοπά είτε σε συσκευασία κυρίως μανταρινιά, από την Κίνα. Η Επιτροπή θέλει να δημοσιεύσει τον, τον εφαρμοστικό κανονισμό με βάση την απόφαση του δικαστηρίου πριν το τέλος, πριν τις αρχές Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε το ζήτημα της, της αναδρομικής ίσπραξης των δασμών. Δίνω το λόγο τώρα στην Γενική Διεύθυνση Trade, που θα έπρεπε να είναι εδώ παρούσα, τον κύριο Γκέρζατ. Παρακαλώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας, αλλά πρέπει να σας πω και κάποιες εξηγήσει Τα μέτρα αυτά για τα μανταρίνια που τα ξέρουμε και ως σατσούμα επιβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 8 αρχικά για να καταλάβουν καλύτερα τους λόγους ε, που το δείς αυτό και για τη σαφήνεια να σας δώσω και τη χρονολογία των γεγονότων στο πλαίσιο αυτό. Καθώς δύο αποφάσεις ε, του δικαστηρίου ακύρωσαν τον κανονισμό του Συμβουλίου του 2008. Η απόφαση της 17ης Δευτέρου 11 το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τον κανονισμό ως προς δύο εξαγωγείς ε, Κίνας από δύο περιοχές, μία από το Γετζιάν και τον δεύτερο από το Γιουμπέι. Ο λόγος ήταν παραβίαση του δικαιώματος της υπεράσπισης. Στις 22 Μαρτίου 2012 ο ίδιος κανονισμός κρίθηκε άκυρος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πλήρως το σύνολό του, διότι σύμφωνα με το δικαστήριο η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη την ε, αναζήτηση αντίστοιχης ε, τιμή σε αντίστοιχη χώρα για να ε, υπολογίσει το τίμημα. Ζήτη, υποχωρούνται τώρα η Επιτροπή να εφαρμόσει την ε, απόφαση του δικαστηρίου και να καλύψει τα κενά που εντόπισε το δικαστήριο. Τούτο γίνεται με μια έρευνα που είναι αρκετά σύνθετη ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης. Επιπλέον, η έρευνα αυτή πρέπει να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια με όλες τις πλευρές και να σέβεται ε, πολύ προσεκτικά τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Εν ολίγης, η προσέγγιση είναι παρόμοια με μια έρευνα anti-dumping που ήθι, όπως ήθιστε που κρατά περίπου τους 15 μήνες. Οι δύο έρευνες που είχαν στόχο να καλύψουν τα προβλήματα που έθεσαν οι δύο αποφάσεις του δικαστηρίου ξεκίνησαν η μία το 2011 και η άλλη το 2012. Η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση εν μέρει ε, ανοίγοντας εκ νέη την έρευνα στις 3, για την πρώτη απόφαση στις 3 Δεκεμβρίου του 2011 και μια δεύτερη προειδοποίηση που ανοίγει εν μέρη την έρευνα μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου του 2012. Κατά τη διάρκεια των ερευνών ήθιστε να μην, ε, ε, ισχύουν τα μέτρα αυτά που σημαίνει ότι οι εισαγωγέ μπορεί να γίνουν χωρί να πληρώνουν ε, δασμού αντι-dumping. Ωστόσο, ο κλάδο υπέβαλε στοιχεία ότι πιθανή επανυποβολή μέτρων θα υπονομευόταν λόγω μαζικών εισαγωγών. Οπότε η Επιτροπή στις 29 Ιουνίου του 2012 δημοσίευσε η Επιτροπή έναν κανονισμό που επιτρέπει εισαγωγέ μετά από καταχώρηση. Ο κανονισμό αυτό επιτρέπει την ίσπραξη των, αναδρομικά την ίσπραξη των δασμών για τρει μήνε σε ορισμένε, ή, εάν πληρούνται ορισμένε ουσιαστικέ προποθέσει. Οι δύο έρευνε ολοκληρώθηκαν, διεξήχθησαν παράλληλα και τα συμπεράσματά του υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2012 σε όλου του ενδιαφερόμενου. Σημειώστε ότι σε αυτό το σύνθετο φάκελο η... χρησιμοποιήθηκε πλήρως η... τα δικαιώματα που αναφέρονται στην νομοθεσία για, την... για το αντι-dumping και οι, οι εγκαλούμενοι χρησιμοποίησαν όλα τα μέτρα που μπορούσαν να του δοθούν. Ζητήθηκαν για παράδειγμα ακροάσεις με τις υπηρεσίες τη Επιτροπής και εποπτεία της ίδιας, παρακολούθηση της ίδιας της ακρόασης. Αυτά τα διαφορετικά βήματα βεβαίως πήραν χρόνο. Ήταν ωστόσο αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία και οι δικονομικοί κανόνες ε, ε, τηρούνταν πλήρως. Η Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη-μέλη μπόρεσε μετά από αυτό να υιοθετήσει στις 28 Ιανουαρίου του 2013 μετά στο Συμβούλιο μια πρόταση κανονισμού που επιβάλλει ε, οι δασμοί στα εν λόγω προϊόντα να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά που αρχικά είχαν καθοριστεί. Το έγγραφο αυτό εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου. Από, το τις 22 Φεβρουαρίου λοιπόν τα μέτρα ε, είναι ενισχύ. Σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα, το ζήτημα θα εξεταστεί προσεκτικά από την Επιτροπή όταν λάβει τα στατιστικά για τις εγωγές σατσούμι μανταρινιών από την Κίνα. Αυτό θα πάρει κάποιες εβδομάδες μετά το δημοσίευση του κανονισμού που επανεπιβάλλει το μέτρο αυτό. Όταν είναι διαθέσιμα πλέον τα στατιστικά θα υποβληθούν τα συμπεράσματα στα μέρη και στα κράτη-μέλη και, ε, και η απόφαση θα ληφθεί από την Επιτροπή μετά από τη διαβούλευση για το θέμα αυτό, ενώ θα υποβληθεί πρόταση και στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά την πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού που επιβάλλει τα συγκεκριμένα μέτρα, σας υπενθυμίζουμε ότι τα μέτρα θα εκπνεύσουν στο τέλος του έτους, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για αναθεώρηση της ε, εκπνοής από τον κλάδο της Ένωσης. Αυτό θα γίνει έξι μήνες τουλάχιστον πριν εκπνεύσουν τα μέτρα, που σημαίνει πριν το τέλος του Ιουνίου του 2013. Επίσης, η νομοθεσία προβλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί έρευνα να αλλάξει το επίπεδο των μέτρων αν αποδειχθεί ότι το επίπεδο του δασμού δεν είναι επαρκές διότι άλλαξε ο βαθμός dumping. Ένα αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί από, από τον κλάδο της Ένωσης αλλά και από τους εξαγωγείς ή εισαγωγείς. Και για τις δύο αυτές δυνατότητες βεβαίως στη φάση αυτή είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε αν ε, θα γίνει θα υποβληθεί αίτημα για αναθεώρηση της εκπνοής ή για αναθεώρηση του επίπεδου δοσμών. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε αγαπητέ εκπρόσωπε της Επιτροπής σας. ξεχίζουμε τη συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτον, να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις ε, εξαιρετικές εξηγήσεις που μας έδωσε. Όπω είπε η Επιτροπή, στι 22 Φεβρουαρίου η Επιτροπή δημοσίευσε τον κανονισμό που επαναφέρει τα μέτρα αντι-dumping για τα μανταρίνια σε κονσέρβα εκ Κίνα ορμόμενα. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω την Επιτροπή που δημοσίευσε τον κανονισμό. Το πρόβλημα είναι ότι το δικαστήριο ακύρωσε την ρήτρα αντι-dumping μέχρι τη, και μέχρι τις 22 Δευτέρου υπήρχε ένα νομικό κενό, που εκμεταλλεύτηκαν οι εισαγωγείς. Αρχές ε, Ιανουάριο και Φεβρουάριο έγιναν μαζικές εισαγωγές μανταρινιών σε κονσέρβα από την Κίνα που είναι αρκετέ για να καλύψουν την κοινωτική αγορά όλο το 2013. Αν δεν υπάρχει αναδομικότητα λοιπόν των μέτρων ε, που δημοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο τουλάχιστον τριών μηνών, η βλάβη στον κλάδο θα έχει ήδη γίνει και θα είναι... δεν θα μπορεί να διορθωθεί και ο κλάδος, όπως είπε η Επιτροπή, τονίζει την ανάγκη και ζητούμε από την Επιτροπή να καταγράφει τις εισαγωγέ. Θεωρούμε ωστόσο ότι μόνο εφαρμόζοντας την ανδρομικότητα από την αρχή της περίοδου θα πετύχει το στόχο να προασπίσει τον ευρωπαϊκό κλάδο και να εισπράττονται οι δασμοί αντι-dumping, που είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Επιπλέον είπε η Κομισιόν ότι περιμένει ακόμα τα στοιχεία. Νομίζω ότι τα στοιχεία υπάρχουν ήδη στα Μητρώα και το γεγονός ότι απλά δημοσιεύτηκε η διόρθωση είναι σαφή, δίνει σαφή εικόνα της κατάστασης. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανάγκη της αναδρομικότητας ε, του κανονισμού δικαιολογείται απόλυτα. Αν περιμένουμε ωστόσο ε, και άλλα στοιχεία θα ζητούσα από την Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί και να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να λύσει το πρόβλημα. Μίλησα και για το μέλλον. Θυμίζω τη σπουδαιότητα του κλάδου και σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασία και την ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα και μετά το 2013 για να διατηρηθεί ο αγροβιομηχανικό ιστός στις παραγωγικές περιοχές. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν οι εργασίε γρήγορα για να υπάρχει ένα νέο κείμενο και για μετά το 2013. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος... Η κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ. Δεν θα, δεν θα μιλήσω πολύ γιατί δεν επαναλάβω αυτά που είπε η συνάδελφος. Να, να εκφράσω τη χαρά μου διότι η Επιτροπή με το που τέθηκε το θέμα για τα μανταρίνια πριν από κάποιες εβδομάδες μέχρι τώρα κατάλαβε τη σοβαρότητα του προβλήματος ε, και τις επιπτώσεις ε, που έχει η έλλειψη ταχύτητας και επιμέλειας από πλευράς Επιτροπής για τους Ισπανούς παραγωγούς και αντέδρασε. Νομίζω ότι το θέμα είναι εθνικό, γιατί βεβαίω η παραγωγή της ποικιλή αυτή είναι καθαρά ισπανική. Αν δεν αναλάβουμε δράση γρήγορα τόσο, διακυβεύεται το μέλλον πολλών ισπανικών οικογενειών που ασχολούνται με, το, με τον κλάδο. Οι αποφάσεις μας λοιπόν επηρεάζουν τους ανθρώπους. Οι εισαγωγέ από Κίνα μόνο μεταξύ Μαρτίου Ιουνίου πέρσι, πέρσι ήταν το ισοδύναμο ολόκληρης της περίοδου. Αν δεν υπάρξει ταχεία αντίδραση από τι και φέτο στην ίδια κατάσταση θα βρεθούμε. Ο κλάδος υποψιάζεται ότι τώρα γίνεται το ίδιο και όταν το υποψιάζεται συνήθως έχουν κάποια στοιχεία. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είμαστε επαρκώς γρήγοροι να, να προστατεύσουμε την ισπανική ευρωπαϊκή παραγωγή παρότι γνωρίζουμε σαφώς ότι υπάρχει αθέμητο εμπόριο που προκύπτει από τις αγωγές αυτές από την Κίνα. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση που έκανε η κυρία Γκαρθία. Τι περιμένει επίση επιτέλους η Επιτροπή για να εφαρμόσει την αδρομικότητα. Είναι αναγκαία για την ε, Ισπανική βιομηχανία. Πέντε επιχειρήσει υπάρχουν στην Ισπανία και οι πέντε μπορεί να χαθούν αν δεν κάνουμε κάτι. Υπάρχουν, θα, θα υποστεί τεράστια βλάβη ο παραγωγικός κλάδο. Σοβαρότατη βλάβη που θα επηρεάζει όχι μόνο τη μεταποίηση, αλλά και την ισορροπία τη αγορά νοπού. Μην ξεχνάτε ότι η μεταποίηση επιτρέπει την εξυγίανση τη παραγωγή νοπού. Επιπλέον, αν τα μέτρα αντι-dumping επεκταθούν μέχρι το Δεκέμβριο φέτο, θα ήταν αναγκαίο να υπάρξει νέα παράταση για να μην υπάρξει αθέμητο ανταγωνισμό τη Κίνα στην κοινωτική αγορά. Ή μήπω σκέφτεται η Επιτροπή ότι θα αλλάξει τον τρόπο εμπορίου τη η Κίνα το Δεκέμβριο ε, ενώ δεν το έκανε ποτέ μέχρι τώρα. Και αντίθετα μάλιστα. Ήταν εξαιρετικά επιθετική. Λοιπόν, νέα παράταση είναι αναγκαία. Χρειάζεται να ξεκινήσει νέα έρευνα από πλευρά Επιτροπή και η αίτηση, το αίτημα των παραγωγών ήδη έχει ξεκινήσει. Περιμένουμε λοιπόν από την Επιτροπή να δράσει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θέλετε μιλήσετε, κύριε της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις ε, που μόλις ακούσαμε ως προς το τι με με αυτά τα μέτρα. Η Ισπανική βιομηχανία δυνατέ να συνεχίσει, τη, να ζητήσει τη συνέχεια των μέτρων ε, καταθέτοντας μια αίτηση ad hoc ε, πριν τον Ιούνιο. Αν το κάνετε αυτό και αν είναι δέοντος αιτιολογημένη η αίτησή σας, θα ανοίξει μια έρευνα και κατά τη διάρκεια της ε, διεξαγωγής της έρευνας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα μέτρα και μετά το πέρας της έρευνας θα ληφθεί απόφαση. Αν ε, θα παραμείνει ενισχύ ή όχι. Σε κάθε περίπτωση σημειώσαμε τις παρατηρήσεις σας. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Έχουμε δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους συναδέλφους. 18-19 Μαρτίου η προσεχής συνεδρίωση. Απόγευμα η πρώτη, από το πρωί η δεύτερη. Χαίρετε.